αυτό στην ημερησία διάταξη. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να υπάρξουν ουσιαστικές επενδύσεις στην Ένωση ε, τα επόμενα χρόνια ξεκίνησε τον προηγούμενο Νοέμβριο, εμείς παίξαμε το ρόλο μας σήμερα υποστηρίζοντας την εκκίνηση εφαρμογής τους. Κάναμε και κάποιες θετικές νομίζω αλλαγές και για το Ευρώπη 2020 όπως επίσης και για το Connect Europe να μην φυγούν. Η Ιρλανδία θα υποστηριχθεί μέσω από τα ταμεία τα κοινοτικά σαν παράδειγμα έχει ήδη κατατεθεί ένα αίτημα για ένα πρόγραμμα κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και έχοντων ανάγκη. Κάποια από τα κέντρα αυτά είναι στο Kildare, στο Galway, στο Westport, στο County Mayor και στο Roscommon. Είναι σημαντικές επενδύσεις όχι μόνο σε υποδομές αλλά στους ανθρώπους τους ίδιους. Ευχαριστώ πολύ. Σντεχόφσκι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ αργά. Γι' αυτό θα είμαι επιγραμματικός. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή συνιστά θρίαμβο όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στην κατάσταση και χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή και συγχαίρω την Επιτροπή Juncker γιατί η σύσταση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα ωφελήσει όχι μόνο τους ετούντε ε, και δικαιούχους, αλλά θα δημιουργήσει μεγάλη προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζήτημα μόνο παρέμεινε αναπάντητο, το θέμα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ ελπίζω να λάβουμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Γιούνκερ. Αυτά και σας εύχομαι καλό βράδυ. Ja sitten äänestysselitykset talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, tilannekatsaus ja haasteet ja edustaja Harkin, olkaa hyvä. Για το δεύτερο τώρα θέμα, η κυρία Χάρκιν η πρώτη ομιλήτρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση γιατί θεωρώ ότι η ευελιξία που υπάρχει στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχική ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευελιξία μέσα στο Σύμφωνο άλλωστε το αναφέρει ήδη. Και θέλω να συνεργαστούμε ε, μαζί με τους Ιρλανδούς Ευρωβουλευτές αλλά και τους λοιπούς συναδελφούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για να υποστηρίξουμε αυτές τις προτάσεις. Έχουμε εγκρίνει με το δημοψήφισμα κανόνες που θα πρέπει να τηρηθούν Γι' αυτό θεωρώ ότι μέσω της έκθεσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν υπάρχει περιθώριο για ευελιξία, γιατί πάνω απ' όλα στο θέμα αυτό χρειάζεται σαφήνεια, χρειάζεται προβλεψιμότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρε, κύριος, η Πρόεδρος και ο κύριος Μπάλτσο. Ο κύριος Μπάλτσο, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τον Οκτώβριο του 2008, ο τότε πρόεδρος ε, Νικολάς Σαρκοζή πρότεινε μία νέα οικονομική διακυβέρνηση. Ουσιαστικά πρότεινε τη δημιουργία ενός υπερκράτους. Άλλαξαν το όνομά του όμως και το αποκάλεσαν οικονομική διακυβέρνηση και όχι ανεξάρτητο οικονομικό φορέα. Αλλά για το ίδιο πράγμα πρόκειται τα κράτη χωρούν ένα μέρος της, κυριαρχία τους, της κυριαρχίας τους για οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συζητούν τους προπολογισμού τους στο Κοινοβούλιο και μάλιστα να προσκαλούν και τους αρμοδίους επιτρόπους για την χρηματοδότηση την κοινοτική στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τα Εθνικά Κοινοβούλια και εξετάζει το σχέδιο προπολογισμού. Και αυτό το κάνει υποτίθεται στο όνομα της δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψήφισε την έκθεση Μπέρες για την οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριος Μαμίνκης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε την έκθεση της συναδελφού Περβάνς Περές. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η κρίση στην Ευρωζώνη έχει πλήξει κράτη. Πολλά. Σε όλη την Ευρώπη, από το 2009 μέχρι το 2011 η Λετωνία ήταν σε πολύ σοβαρή κρίση, ακόμα δεν την έχει ξεπεράσει και στο βαθμό που την ξεπέρασε δεν την ξεπέρασε χάρη στις βοήθειες, στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χάρη στις προσπάθειες του λετωνικού λαού, ο οποίος δέχθηκε τεράστιες περικοπές σε συντάξεις και μισθούς αλλά ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοιες πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, να βρούμε συμβαστικές λύσεις μεταξύ όλων των πλευρών. Και γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση της Περβάνος Περές, γιατί είναι μια συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι ολοκληρώνονται